Οι Ισπανικές Αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή της κυρία Τάνια Γκοντζάλιας Πένιας ε, από 10 Σεπτεμβρίου 2014. Η κυρία Γκοντζάλιας Πένιας ε, αντικαθιστά τον Κάρλος Χιμένες Μιλαρέχου. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 ε, της πράξης για την άμεση εκλογή των Ευρωβουλευτών και το άρθρο 4 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση τη εκλογή τη κυρία Γκονζάλης Πένια από 11 Σεπτεμβρίου 2014. Καλώς ορίζουμε τη συνάδελφο και να σα υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου εφόσον δεν ε, υπάρχει κάποια